l'encadrement réglementaire pour les entreprises, la confiance des consommateurs et la gouvernance du marché unique. Thank you very much. Three very clear priorities there. Minister, if I could turn to you now. What do you see as the key challenges that lie ahead? Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι που χρειάζεται είναι η ευάθυνση της ενιαίας αγοράς. Και χρειάζεται βεβαίω εδώ να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, διότι η ευάθυνση της ενιαίας αγοράς θα βοηθήσει πρώτα-πρώτα να ε, προωθηθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση, ε, ειδικά στις, ε, ιδίως στις ψηφιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις δικτύου. για, να προ, για να προωθηθεί αυτό χρειάζεται πρώτα-πρώτα να κινηθούμε πιο γρήγορα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας πράξης αγορά 1 και να βάλουμε το συντομότερο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την υλοποίηση τη ενιαία πράξη αγορά 2. Ε, με αυτή την ευκαιρία, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Μισελ Μπαρνιέ γιατί, ε, για την ανακοίνωση τη Επιτροπή ε, η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα στι 12 του Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο και είναι σε ένα τομέα που πρέπει να δουλέψουμε εντατικά. Η ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά θα βοηθήσει ακριβώ ε, το να λειτουργήσουν πιο ανταγωνιστικά επιχειρήσει ε, στην Ευρώπη και αυτό είναι καλό και για την οικονομία αλλά και για του πολίτε. Το δεύτερο είναι χρειάζεται ταχεία πρόοδο σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία τη ψηφιακή ενιαία αγορά που πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το 2015. Είναι, ε, αυτή η διαδικασία είναι κάτι που θα προσδώσει ένα νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία σε έναν τομέα πολύ σημαντικό. Το τρίτο είναι η η ολοκλήρωση της ε, αγοράς ενέργειας, η οποία τέθηκε ως στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Πρέπει να, να είμαστε συνεπείς σε αυτές τις ε, προθεσμίες και βεβαίως να διασφαλίσουμε ε, ότι μετά την ολοκλήρωση το 2014 της αγοράς ενέργειας κανένα κράτος στην Ευρώπη δεν θα είναι απομονωμένο από τα ενεργειακά δίκτυα. Άρα θεωρώ αυτές τις τρεις σημαντικές προκλήσεις ε, για την ίδια την ε, ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, για την ίδια την οικονομία της Ευρώπης, για να προσδώσουμε νέα δυναμισμό στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.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 It's not always easy. Do we need more? Do you feel that the single market is getting uh the political will behind it from the member states that it really needs? Ναι, να πω ότι βεβαίω ε, η πολιτική βούληση υπάρχει ε, για να προχωρήσει και να εμβαθυνθεί η ενιαία αγορά. Όμω, ε, εγώ θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα από αυτήν την παρουσία που είχαμε. Φαίνεται ότι με τι απαντήσει οι πολίτε πιστεύουν στην ενιαία αγορά αυτό που χρειάζεται και στην ευβάθυνσή τη, σαν απάντηση και στην κρίση. Ε, Εμεί τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα, θεωρώ ότι ε, οι, οι, αναλύσει που κάνουμε κινούνται από όλου στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα λόγω τη οικονομική κρίση κινδύνου για τα επιδέγματα 20 χρόνων ενιαία αγορά, και αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Υπάρχει και ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό που ενδεχομένω δημιουργά προβλήματα. Υπάρχουν νέα φαινόμενα, κλιματικές αλλαγές, τεχνολογική ε, αναβάθμιση ε, και εδώ πρέπει ακριβώς να δουλέψουμε για να, ε, να απαιτούν όλα αυτά τα νέα δεδομένα, νέες απαντήσεις, νέους κανόνες. τώρα άκουγα που είπε και ο Μισελ και αναφέρθηκε και εσύ κυρία Τέλης για τα θέματα της του e-signature, e-commerce μπορώ να πω, e-learning Όλα αυτά είναι νέα φαινομένα που πρέπει εμεί να δημιουργήσουμε του κανόνε σήμερα, όχι αύριο. Και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Εκείνο που χρειάζεται όμω είναι όλοι να δουλέψουμε συλλογικά. Αλλά θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα στην αρχική μου παρέμβαση. Χρειάζεται να κινηθούμε πιο γρήγορα. Αναφέρθηκε ο Μισελ για πολλά ζητήματα yeah. που έχουμε μπροστά μα. Είτε για τι οδηγίε ATR, ε OTR, για τι δημόσιε συμβάσει, για τα επαγγελματικά προσόντα που θα βοηθήσουν στην κινητικότητα. Όμω διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες. Ενώ είχαμε, είχε τεθεί ο στόχο ότι μέχρι το τέλο τέλος του 2012 θα ολοκληρώσουμε, θα ολοκληρώναμε την ενιαία ένα, τότε ε, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Ε, τα συζητήσαμε στο τελευταίο συμβούλιο την περασμένη ε, Πέμπτη στο Λουξεμβούργο. Ε, από τη δική μας πλευρά ως Προεδρία θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ολοκληρώσουμε όσο περισσότερους φαγγέλους ε, υπάρχουν και να ξεκινήσει και η συζήτηση όπως ξεκίνησε για την ενιαία αγορά 2. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Η κρίση ε, έχει μια χρονική διάρκεια ε, ε, σε και αγκαλιάζει όλο ένα και περισσότερα κράτη και πολίτες στην Ευρώπη. Χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις σήμερα και να δώσουμε απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.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 Ε, αυτό είναι σωστό πως ο, ο πολίτης θα υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα και των πολιτών βεβαίως και των επιχειρήσεων σε όλους τους αυτούς τους κανόνες. Αυτό που συζητούμε τώρα πρώτα-πρώτα είναι να απλοποιήσουμε τους κανόνες, να τους κάνουμε πιο προσιτούς, να αποφορτώσουμε ε, και διοικητικό ε, άχθος από τις ε, επιχειρήσεις, αλλά να διευκολύνουμε και τον πολίτη. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αναφέρθηκα προηγουμένω ε, και στι ε, εναλλακτικέ ε, μεθόδου επίλυση διαφορών του καταναλωτή. Πώ διευκολύνουμε το καταναλωτή. Ε, το τρίτο ζήτημα είναι το ότι ε, προηγουμένω δημιουργήσαμε νέα κέντρα εξυπηρέτηση. Αυτά πρέπει να διευρύνουμε την εφαρμογή του, να μπορεί ο πολίτη να φτάσει πιο κοντά στα προϊόντα μέσα από την αγορά και να έχει περισσότερη ε, διαφάνεια επίση στι ε, διαδικασίε μα, ειδικότερα στι υπηρεσίε και για να μην αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, γιατί μιλούμε για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και όμω εδώ υπάρχει πρόβλημα πώ θα μπορέσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να επιβιώσουν μέσα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική κρίση. Άρα, συζητούμε του κανόνε, είμαστε μπροστά σε νέε προκλήσει και νέε ανάγκε. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένω για να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και να φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να μην αναφέρθηκε στη συζήτηση. Εδώ και 20 χρόνια προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ε, το κέντρο ε, για τη ε, θέματα της εύρης τεχνίας. Μιλούμε για νέες καινοτομίες, νέα προϊόντα και ακόμα δεν ολοκληρώσαμε αυτό το ζήτημα και ελπίζω να το ολοκληρώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει δυνατότητες ε, και ε, σε πολλές επιχειρήσεις να πλασάρουν νέα προϊόντα στην αγορά και πρέπει ακριβώς για να λειτουργήσουμε στην κοινωνία να δημιουργήσουμε ε, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που ανάφερα προηγουμένως. Thank you. Thank you very much. So, to the yes, please, Vladimir, talk from you. Uh, uh, thank you, Jackie, very much for this question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 Thank you for giving me the floor. I would like to address the House in Greek, please. Λέγομαι Γιώργος Σιλιόπουλος, είμαι φοιτητής, εκπροσωπώ και εγώ τη γενιά του 1992 και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σύγχρονη πρόκληση της ενίας ευρωπαϊκής αγοράς που είναι ενεργεία. ανεργία. Ε, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα είναι 23,6% περίπου και 50% ειδικά στην ε, ομάδα των νέων. Ε, εγώ για να βοηθήσω τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν κάποια δουλειά δημιούργησα μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα η οποία βοηθάει στη συγγραφή, στη δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος. Ε, ωστόσο, για να βρεις κάποια εργασία θα πρέπει να υπάρχει εργασία, θα πρέπει να υπάρχει προσφορά εργασίας. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, να αλλάξει στις δομές και στη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες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 and uh, I'll take the advantage to follow to my mother tongue, the Greek. So, ε, θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει περισσότερα για τα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς και τις επιχειρήσεις των μηχανικών ε, εάν ε, είχε δοθεί ο λόγος στον κύριο Lars Bitoft της European Federation of National Engineering Associations ο οποίος από ό,τι έμαθα δεν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως να είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω το εξή ότι εμείς οι μηχανικοί και οι επιχειρήσεις των μηχανικών ε, έχουμε βρει τον τρόπο να κινούμαστε στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, υπάρχουν μερικά εμπόδια ακόμα. Συζητάμε πάρα πολλά χρόνια την οδηγία, την PQD, Professional Qualifications Directive, αλλά νομίζω μαζί με τους ε, άλλους οργανισμούς, τη ΦΕΑΝΗ και εμάς, ότι θα μπορέσουμε να τους λύσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν των μηχανικών, το πρόβλημα των τεχνικών υπηρεσιών ε, είναι ένα άλλο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πόροι για αυτό που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν οι Ευρωπαίοι και είναι υποδομές. Τα ITs είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, αλλά είναι στα χέρια των Αμερικάνων, στα χέρια των Ινδών, στα χέρια των Κινέζων. Τι λοιπόν μπορεί να γίνει με το ε,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 Ναι, ε, πρώτα πρώτα να, ε, να πω μερικά σχόλια ξεκινώντα από αυτό για κάποιε παρατηρήσει. Ε, η συμπατριώτησα μου αναφέρθηκε για, ακριβώς για, για το επιχειρηματικό πνεύμα. Ε, στο άτυπο συμβούλιο που ξεκίνησε η Κυπριακή Προεδρία ε, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην Κύπρο, κύριο θέμα ήταν η επιχειρηματικότητα η νεανική επιχειρηματικότητα, η γενική επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Ανταλλάξαμε, και μάλιστα, ανταλλάξαμε καλές ιδέες. Ε, είχαμε μάλιστα ε, ε, είχαμε συμμετάσχοντες και ομιλητέ στο συνέδριο ανθρώπου και από την επιστήμη και από την παραγωγή. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση θα μας βοηθήσει να οδηγηθούμε ώστε στο επόμενο συμβούλιο που θα γίνει τον Δεκέμβριο εδώ στις Βρυξέλλες να βγάλουμε συμπεράσματα γι' αυτό. Ε, και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλέ ιδέε. Ε, δηλαδή, όμω εκεί που πρέπει να προσεγγίσουμε πάντοτε και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε καλέ ιδέε. Διαμορφώνουμε και με ανακοινώσει τη Επιτροπή και μετά με συμπεράσματα του Συμβουλίου αυτέ τι πολιτικέ. Εκεί που είναι το δύσκολο είναι αυτές τις πολιτικές που χαράζουμε να τις μεταφέρουμε στην πράξη. Να μετατραπούν δηλαδή σε κανονισμού και νομοθεσίε που θα βαστούν πολιτικέ. Εδώ είναι η μακρόχρονη διαδικασία. Εδώ είναι που δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, ε, εδώ θέλουμε ε, για να εφαρμόσουμε καινοτομία χρειαζόμαστε και νέου κανόνε, αλλά χρειαζόμαστε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά δεν είναι αρκετά. Το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, επειδή αναφέρθηκε από τον ε, συνάδελφο το λέω συνάδελφο και εγώ είμαι μηχανικός από την Ελλάδα, ε, να πω πριν από για τα θέματα των επαγγελματικών προσόντων που είναι ένα από τους δύσκολους φακέλους που διαχειριζόμαστε τώρα. Ε, και έχουμε διαφωνίες μεταξύ των μελών, ενώ όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διευκολύνουμε την κινητικότητα και είναι βασικό για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων να, ε, να, να ολοκληρώσουμε αυτόν τον νομοθετικό φάκελο. Εν τούτης ακόμα υπάρχουν δυσκολίες και να πω ότι το τελευταίο, ότι στο τελευταίο συμβούλιο ε, που αναφέρθηκα προηγουμένω ε, στο Λουξεμβούργο, ε, κύριο θέμα μα δεν ήταν η νέα αγορά. Κύριο θέμα μα ήταν η νέα βιομηχανική πολιτική. Και είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Μιλούμε για ανταγωνισμό, μιλούμε για νέα κέντρα στην περιφέρεια που μα ανταγωνίζονται, αλλά χρειαζόμαστε νέε βιομηχανικέ πολιτικέ σε πολλά ζητήματα. Είναι θετικό το γεγονό ότι κατορθώσαμε μετά από πολλή συζήτηση να έχουμε συμπεράσματα για τα CATS, ε, τη ε, μηχανολογία τεχνολογία και την καινοτομία στι πρώτε ύλε. Ε, αναφέρομαι σε δύο τομεί που ένα τομεί αντιμετωπίζουμε ω ό,τι αφορά τα ΚΕΤ μεγάλων ανταγωνισμών από επιχειρήσει από την περιφέρεια και στον άλλο τομέα που αναφέρομαι στι πρώτε ύλε που η Ευρώπη εν πολύ σε μεγάλο βαθμό είναι εξαρτημένη από εισαγωγέ. Άρα μιλούμε για νέου τομεί που θα βοηθήσουν και τη βιομηχανία αλλά θα βοηθήσουν να γίνει πιο ανταγωνιστική αλλά θα βοηθήσουν και τις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 Θα ξεκινήσω από εκεί που άρχισα στην αρχή, ότι αυτό που χρειάζεται είναι σήμερα εμβάθυνση τη ε, ενιαία αγορά. Και εμβάθυνση πρώτα και κύρια σημαίνει καλύτερη διακυβέρνηση. Απλοποίηση των διαδικασιών, διαφάνεια, και όταν λέω διαφάνεια, αυτό που χρειάζεται σήμερα πάνω απ' όλα είναι να υπάρξει διαφάνεια στου χρηματοπιστωτικού κανόνε, ε, ασφάλεια στα προϊόντα και, και βεβαίω στα τρόφιμα, ε, διευκόλυνση της διακίνησης, ε, ανοιχτές ανταγωνιστικές και τεχνολογικά αναπτυγμένες τηλεπικοινωνίες, ασφαλής ανταγωνιστική και αποτελεσματική ενεργειακή αγορά, διότι ένας από τους σημαντικούς ε, τομείς, ε, και ε, ε, θεωρώ ότι αυτά όλα μπορούν να εκφραστούν με τους νέους κανόνες και διευκόλυνση βεβαίω να εισάγουμε νέα καινοτόμα προϊόντα νέε καινοτόμε διαδικασίε, να διευκολύνουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία για την εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην αγορά. Έτσι θα δώσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον πολίτη, θα δώσουμε δυνατότητε ανάπτυξη ε, και δημιουργία ε, πολλών θέσεων εργασία. Thank you very much indeed, Minister. And before we close, I'd just like to read you one more tweet, uh, because I think this is a rather marvellous tweet. It's from Emmanuel van Praag, and he simply says,